Okay, dear colleagues, uh, let's start our... Ας ε, ξεκινήσουμε τη συνεδρία της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου μετά την συνεδρίαση με την ΕΜΚΟ. Σας, ε, θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας στην ακρόαση. Με χαρά μου είδα πολλά μέλη της ε, δική μα επιτροπή ενώ λίγα μέλη τη επιτροπή ΣΥΜΚΟ. Κάναμε λοιπόν πολύ καλή παρουσία και με γέμισε περηφάνεια. Σημείο 2. Έγκριση τη ημερήσια διάταξη. Δεν υπάρχει κανένα αίτημα τροποποίησης της, οπότε υιοθετείτε. Σημείο 3 έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης της 14ης και 15ης Μαρτίου. Τα πρακτικά θα υιοθετηθούν στο τέλος συνεδρίασης εκτός και αν μέχρι τότε έχει φτάσει κάποιο σχόλιο στα χέρια μας. Σημείο 4. Ανακοινώσεις του Πρόεδρου. Θα σας υπενθυμίσω ως συνήθως ότι η συνεδρία μεταδίδεται στο διαδίκτυο και αυτοί που μας βλέπουν από το Τάλινε, από τη Λισαβόνα, από το Λονδίνο, το Άμστερνταμ και αλλού θα προσέχουν σίγουρα τα όσα λέμε πολύ προσεκτικά. για τις ε, διαπραγματεύσεις. Ο επόμενος γύρος θα ξεκινήσει στις 25 ε, Απριλίου στη Νέα Υόρκη για την TTIP. Θα είναι παρούσα και η Σεσίλια Μάλστρομ για να επιταχύνουμε τις διαπραγματεύσεις. Θα δούμε. Σημείο 5. Κατάσταση των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων του τριμερούς διαλόγου. Ε, δεν έχουμε τίποτα καινούριο σε σχέση με τα ε, ορυκτά. Ε, ε στατιστικά εξαγωγικού εμπορίου, εκεί έχουμε κάποια νέα. Πριν από 1,5 χρόνο ε, ο κανονισμός είχε, ήταν στο Συμβούλιο, έφτασε στο Συμβούλιο, αλλά το Συμβούλιο δεν ήταν έτοιμο να δεχτεί το συμβιβασμό. εξαιτία της ε, χρήσης των εφαρμοστικών ε, και κατευσιόδότηση πράξεων, καθώς επίσης και με τις προσκλήσεις ε, εμπειρογνωμόνων από πλευρά ε, Συμβολίου και κομισιών στην ομάδα εμπειρογνωμόνων. Ε, οπότε παρόλο ότι οι διαπραγματεύσει έχουν ολοκληρωθεί στον τριμερή διάλογο, το θέμα εκκρεμεί. Βρίσκεται στο νέφος. Μετά την διοργανική συμφωνία που ολοκληρώθηκε πριν από μερικές εβδομάδες, εισάγαμε στοιχεία αυτής της συμφωνίας στον κανονισμό, οπότε οι διαφορές πλέον έχουν ε, επιληθεί, έχουν εξομαλυνθεί και μπορούμε να ψηφίσουμε αύριο. Περνάμε στο σημείο 6. Προετοιμασία της ε, μετεκλογικής αναθεώρησης του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου Ε, ο κ. Μπέγκε είναι ο συντάκτη νομοδότηση. Του δίνω το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, στην αρμόδια την Επιτροπή προπολογισμών η Ιζαμπέλ Τοβά και ο Γιάννο Όλμπριχτ είναι συνεισηγητέ. Θα κάνω μια σύντομη παρουσίαση σήμερα παρά το ότι αυτά που έχουμε ενώπιον μας ώψη τη αναθεώρηση του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου θα δημιουργήσουν πολλές δυσχέρειες. Πρέπει να είναι σαφές και αυτό θέλω να αποστείλω ως μήνυμα σαφές προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Εάν δεν επιτύχουμε να υπάρξει συμφωνία για ορισμένα βασικά σημεία του προπολογισμού, των πολιετών προοπτικών δηλαδή για το 14-20, εάν δεν το επιτύχουμε, τότε κάθε χρόνο η διαδικασία έγκρισης ε, του προπολογισμού θα είναι πρωτάκουστη και όσον αφορά τις διχογνωμίες και όσον αφορά τη δυνατότητα ο προπολογισμός να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις. Τα τελευταία, τους τελευταίους μήνες είχαμε την κρίση των προσφύγων, είχαμε γι' αυτό διάφορες αναδιατάξεις στον προπολογισμό τόσο μεγάλες που δεν τις έχω ξαναδεί στα 24 χρόνια που είμαι στον προπολογισμό. Έχουμε ναι, 9,2 δις που εγκρίθηκαν με fast track διαδικασία για το 15 και το 16 τον Οκτώβριο. Επίσης θυμίζω ότι μετά από δυσχερείς διαπραγματεύσεις με την Ιρλανδική Προεδρία που παραλίγο να αποτύχουν γιατί υπήρχε πολύ μεγάλη ξεροκεφαλιά και επειδή είχε υπάρξει διαστρέβλωση της παρουσίασης στην κοινή γνώμη του τι είχε συμβεί επιτύχαμε να υπάρξει περισσότερη ευελιξία στη διαδικασία έγκρισης του προπολογισμού για να αξιοποιούμε περιθώρια και ούτως ώστε τα ανώτατα όρια για πληρωμές και υποχρεώσεις παρόλα αυτά να διατηρηθούν δηλαδή τα 960 και τα 908 δις, γιατί από την αρχή ήταν σαφές ότι λόγω της καθυστέρησης των διαπραγματεύσεων για την νομική βάση των πολιετών προγραμμάτων θα υπήρχε γενικότερη καθυστέρηση. Και ήταν σαφές ότι θα αντιμετωπίζαμε και πάλι την κατάσταση λοιπόν που έχουμε και σε άλλες ε, μεσοπρόθεσμε δημοσιονομικέ διαδικασίε, ότι κάποια ποσά καταπίπτουν και πρέπει να διαγραφούν. Αυτό που είναι ενδιαφέρον που αφορά την εργασία μας εδώ είναι ότι αυτό το πρόβλημα δεν το αντιμετωπίζουμε μόνο στις διαθροτικές πολιτικές αλλά τα τελευταία χρόνια όλο και πιο συχνά διαπιστώνουμε ότι ορισμένα μέσα εξωτερικής πολιτικής δεν μπορούν να υλοποιηθούν πλήρως. Αυτό σε μεγάλο βαθμό έχει να κάνει με την κατάσταση στις χώρες ε, όπου θέλουμε να δαπανηθούν τα χρήματα αυτά ή με τις χώρες όπου θέλουμε να υπάρξουν εταιρικέ σχέσεις για να συμβάλλουμε στη μεσοπρόθεσμη σταθεροποίηση των κοινωνιών. Προκύπτουν εκεί γεγονότα που δεν μας επιτρέπουν να εφαρμόσουμε αυτά τα οποία θα θέλαμε να κάνουμε. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να είναι σαφές σε όλους μας ότι αντιμετωπίζουμε προκλήσεις σε αυτή τη συγκυρία και ότι οι καταστάσεις ε, στις ε, πάνε στις κατηγορίες 3 και 4 σημαίνει ότι πρέπει να ληφθούν αποφάσεις. <clears throat> Και όχι μόνο, για παράδειγμα, όταν συζητάμε για το προσωπικό της Europol και της Frontex, όπου, για παράδειγμα, το περασμένο καλοκαίρι ενώ ήμασταν εν μέσω της κρίσεως, ε, το Συμβούλιο αρνήθηκε να δράσει εγκαίρως. Το βασικό καθήκον μας, πέρα από πολλά άλλα, πρέπει να είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε τις καταστάσεις ε, στις γειτονικές μας περιοχές στην Εγγύς και Μέση Ανατολή και στην Αφρική, ούτως ώστε να συμβάλλουμε στην διαρκή σταθεροποίηση για να μην απειλούμεθα συνεχώς από ε, κράτη, από κράτη που έχουν καταρρεύσει. Και εδώ τίθεται το θέμα πώς θα ε, ενταχθεί και η εμπορική πολιτική σε αυτή την προσπάθεια, γιατί είναι αποφασιστική σημασία. Ε, στην κατηγορία 4 έχω αναφέρει αρκετά στην ε, γνωμοδότησή μου. Έχω αναφερθεί στην απελπισμένη προσπάθεια της Κομισιόν με πολλή δημιουργικότητα όσοι επιτρέπουν οι κανόνες του προπολογισμού να αιτιολογήσει τη δαπάνηση ποσών εκτός του προπολογισμού στην ε, συνάντηση κορφής τη ε, Βαλέτα προτάθηκαν 1,5 δί για τη Βόρεια Αφρική από υπάρχοντες γραμμέ του υπερπολογισμού, από τα υπάρχοντα μέσα για την ανάπτυξη και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο ανάπτυξη. Εγώ νομίζω ότι πάντα πρέπει να δούμε πού μπορούμε να κάνουμε αναδιατάξεις γιατί ίσως να προκύψουν προτεραιότητες διαφορετικές από αυτά που είχαμε αποφασίσει και λόγω αυτής της αναδιάταξης καταφέραμε από τα προγράμματα γειτονίας να κανουμε αναδιαταξει γιατι ισω να προκυψουν προτεραιοτητε διαφορετικε απο αυτα που ειχαμε αποφασισει και λογω αυτη τη αναδιαταξη καταφεραμε απο τα προγραμματα γειτονια να βρουμε 500 εκατομμύρια περιμένοντας ότι τα κράτη-μέλη επίσης ε, θα μας έδιναν 1,5, ε, ε, άλλο 1,5 εκατομμύριο εκτός του προϋπολογισμού. Αυτή η διαδικασία επιτρέπεται με βάση το δημοσιονομικό κανονισμό, αλλά γιατί το αναφέρω τόσο πολύ. Γιατί διαπιστώσαμε ότι από ό,τι ξέρω μέχρι σήμερα τα κράτη-μέλη δεν έχουν δώσει αναταμείο ούτε καν 100 εκατομμύρια. Άρα ε, όταν με αυτόν τον τρόπο με διακυβερνητική μέθοδο προσπαθούμε να λύσουμε τα προβλήματα αυτής της κατηγορίας τελικά δεν κάνουμε τίποτα. Ε, υπάρχουν ε, χώρες που μας δίνουν ε, 3 εκατομμύρια και αυτά μένουν στην ε, Διοικητική Επιτροπή, στο Steering Board και αρκούνται σε αυτά. Γι' αυτό τονίζω ιδιαίτερα επικριτικά ότι μπορούμε να εγκρίνουμε τέτοιε λύσει μόνο εάν υπάρχει τεράστια ανάγκη επίγουσας ε, δράσης και δεν θα πρέπει να ε, χρησιμοποιούνται τέτοιε μέθοδοι χρηματοδότηση εκτό προπολογισμού που σημαίνουν και εκτό ελέγχου και έγκριση του προπολογισμού του Κοινοβουλίου. Γι' αυτό στα πλαίσια τη αναθεώρηση πρέπει να πούμε τι αναθεώρηση θέλουμε. Θα επιτρέψουμε τέτοιες λύσεις. Μακροπρόθεσμα κάτι τέτοιο θα έφυγε την κοινοβουλευτική πλευρά τη έγκριση του προπολογισμού. Και ορισμένοι λένε ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε πολύ πιο εύκολα να εγκρίνουμε και να δαπανίσουμε αυτά τα ποσά εκτό τη ε, δημοσιονομική διαδικασία. Τότε πρέπει να πούμε, τι πράγματα είναι αυτά. Εδώ παραβιάζουμε τον δημοσιονομικό κανονισμό. Είναι λοιπόν πολύ περίπλοκη αυτή η κατάσταση, πρέπει λοιπόν με μεγάλη προσοχή να την παρακολουθήσουμε. Και φυσικά το θέμα πώς μπορούμε με περισσότερη ευελιξία να αντιμετωπίσουμε νέες προκλήσεις είναι σημαντικό βέβαια. Αλλά εμείς πρέπει να πούμε ότι πρέπει να έχουμε επαρκείς ε, πιστώσεις για να αντιμετωπίσουμε και να εκπληρώσουμε τους ε, εμπορικούς στόχους της πολιτικής μας και για να συμβάλλουμε στη σταθερότητα, την ανάπτυξη και την απασχόληση και σε εμά και στις γειτονικές μας χώρες. Το συνδέω και με αυτό που είπε ο συνάδελφος Σούστερ για το πώς αποτιμούμε τη χρήση των υπαρχόντων μέσων. Ε, πρέπει να μας πει περισσότερο από αυτού η Κομισιόν. Και στο κείμενό μου θα κάνω κάποιες αλλαγές για να τεθεί το θέμα της αξιολόγησης των υπαρχόντων μηχανισμών και μέσων. Δεν θα πρέπει να μα πούνε οι υπηρεσίε τη Κομισιόν ότι δεν έχουν λεφτά για να το κάνουν αυτό, γιατί ορισμένε φορέ μα το λένε αυτό. Γιατί ορισμένε φορέ στην ουσία είναι πρόσχημα αυτό. Κατόπιν αναφέρομαι στην ε, μεταναστευτική και προσφυγική κρίση, τι πρόκληση έχουμε ενώπιόν μα, ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τα αίτια αυτή τη κρίση. και ότι η εμπορική πολιτική πρέπει να συμμετάσχει σε αυτή την προσπάθεια. Αναφέρω τη στήριξή μας ε, για την ε, ε, διεθνοποίηση του θέματος της στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τη χρήση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων σε σχέση με την εξωτερική πολιτική για να μειώσουμε τους κινδύνους για τα δάνεια που δίνει η Ένωση προς τρίτες χώρες. Και αναφέρομαι επίσης και στα μακροχρηματοδοτικά προβλήματα και τα, τους πόρους που πρέπει να έχουμε στην κατηγορία 5. Να ελέγξουμε τις εμπορικές συμφωνίες, για να μπορέσουμε να ελέγξουμε τις εμπορικές συμφωνίες και να δούμε πώς μπορούμε να τροποποιήσουμε αυτές τις συμφωνίες. Δυστυχώς, δεν έχουμε δυνατότητα που είχαμε πριν από τη Λισαβόνα να καθορίσουμε ε, μονομερώς ε, αποθεματικά στον προπολογισμό. Ορισμένε φορές ακόμη και το κόστος ταξιδιού των επιτρόπων το είχαμε βάλει στο ε, αποθεματικό αυτό. Αλλά αυτό μπορεί να δημιούργησε ανησυχίες, αλλά έχει αποτέλεσμα ότι επιτύχαμε αυτά που θέλαμε. Οπότε πρέπει να σκεφτούμε πώς μπορούμε να επανέλθουμε σε τέτοια μέσα όταν θα συζητήσουμε με το Συμβούλιο τα θέματα αυτά, ούτω ώστε να αντιμετωπίσουμε σοβαρά σοβαρότερα από ότι μέχρι στιγμής αυτά τα προβλήματα. Αυτά ήθελα να πω κύριε Πρόεδρε για την προετοιμασία των διαπραγματεύσεων, για την αναθεώρηση των πολιετών δημοσιονομικών προοπτικών που θα είναι σίγουρα ιδιαίτερα δυσχερής αλλά πρέπει πολύ ε, αποφασιστικά να θέσουμε τις προτεραιότητές μας αλλιώς η δημοσιονομική πολιτική και αυτά που αναμένουμε από αυτήν ε, για τα επόμενα χρόνια απλά και μόνο θα αποτύχει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και ο Πρόεδρος για αυτήν την αναλυτική παρουσίαση. Να στραφώ τώρα προς τους σκιώδεις ή μα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κύριε Πρόεδρε, να συγχαρώ τον ε, συντάκτη της νομοδότησης για το σχέδιο γνωμοδότησης το οποίο μας υπέβαλε και να πω ότι οι σοσιαλιστές θα συνεργαστούν και να σας πω ότι θα υποβάλουμε και τροπολογίες προκειμένου να προσπαθήσουμε να συμπληρώσουμε με κάποια θέματα και να μπορέσουμε, ελπίζω, να τα υποστηρίξουμε όλοι. Δύο σχόλια. Ένα γενικό για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε σε μια μεταρρύθμιση των ίδιων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να μπορέσουμε να διαθέτουμε τα απαραίτητα ποσά για να αντιμετωπίσουμε τις ε, ανάγκες που έχουμε σε δαπάνες και φυσικά να βοηθήσουμε στην επίλυση του προβλήματος των πληρωμών που αντί να μειώνονται αυξάνονται όλο ένα και περισσότερο. Επίσης, να διασφαλίσουμε και τον δημοκρατικό έλεγχο του Κοινοβουλίου στον έλεγχο των πόρων που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, κάποιοι εξ αυτών, όπως είπε και ο εισηγητής, είναι πέραν του προϋπολογισμού, όπως ο μηχανισμός για τη βοήθεια ε, στους πρόσφυγες. Πρέπει λοιπόν το Κοινοβούλιο να είναι σε θέση να ελέγξει όλα τα χρηματοοικονομικά μέσα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όσον αφορά τα όσα μας αναλογούν εμάς ως Επιτροπή, είναι ουσιαστικό να βελτιώσουμε τους πόρους και την αποτελεσματικότητα στις μεθόδους αξιολόγησης και στις ε, εκ των προτέρων και κυρίως εκ των υστέρων εκτιμής επιπτώσεων. Θα πρέπει να έχουμε πολύ πιο αναλυτικό έλεγχο του πώς εξελίσσονται όλα όσα έχουν συμφωνηθεί και κυρίως να δημοσιοποιούνται οι πληροφορίες και οι δυνατότητες που προσφέρονται από τις νέες συμφωνίες, ώστε όλοι όσοι μπορούν να υποβαλληθούν, να υποφεληθούν και να μην ε, ε, χαθούν οι ευκαιρία επειδή δεν γνωρίζουν τι περιλαμβάνουν. Επίσης, ε, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να αναφερθούμε και σε μελέτες επιπτώσεων για τα πιθανά μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να ληφθούν για να βοηθήσουμε τρίτες χώρες σε κατεπίγουσες περιπτώσεις, αλλά να ξέρουμε και τι συνέπειες μπορούμε να έχουμε και στους ευρωπαϊκούς τομείς και ή δυνατόν να προσαρμόσουμε και τα μέτρα στις περιπτώσεις αυτές. Επίσης, να επιμείνουμε στην απαραίτητη μεταρρύθμιση του Ταμείου Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση. Πρέπει να έχει περισσότερου πόρου και να είναι λιγότερο περιορισμένη η δυνατότητα πρόσβαση στο Ταμείο. Οι μικρομεσαίε επιχειρήσει που πλήττονται από την παγκοσμιοποίηση δεν πρέπει να αποκλείονται, γιατί ε, είχαμε θέσει ένα ανώτατο όριο και δεν καλύπτονται. Πρέπει λοιπόν να μπορέσουμε να συνεργαστούμε και να έχουμε ένα πλήρε έγγραφο. Αυτά από πλευρά μου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον εισηγητή που μας παρουσίασε τις σκέψεις του, που συμφωνώ μαζί του. Ε, νομίζω ότι είναι πολύ προβληματική η κατάσταση. Έχουμε ένα προπολογισμό χωρίς πόρους, ένα προπολογισμό χωρίς αξιοπιστία και γι' αυτό είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό πρόβλημα. Υπάρχουν πολλέ ερωτήσει που μπορούμε να θέσουμε για τον προπολογισμό, για τι δαπάνε που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση υπό την έννοια των επιδοτήσεων αντί να κάνει επενδύσει στην οικονομία του 21ου αιώνα. Βέβαια, είναι πολύ ευρία η συζήτηση για να γίνει εδώ στην Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου. Ε, επίσης, θεωρώ ότι πρέπει να εξετάσουμε το εμπόριο ως τμήμα των μέσων που θα μπορούσε να έχει στη διάθεσή της Ευρωπαϊκή Ένωσης εξωτερικής της δράσης και χαίρομαι για τα σχόλια που έγιναν για την έλλειψη αξιοπιστίας και τη δημιουργική χρήση του προϋπολογισμού η οποία υποσκάπτει και την ε, υπόσχεση της ε, εφαρμογής της αρχής για περισσότερα για περισσότερα. Δηλαδή, να υπάρχει μεγαλύτερη πρόσβαση στις αγορές, για παράδειγμα, για μειονότητες, καλύτερες ε, δράσεις και συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οποιαδήποτε κίνηση κάνουμε στην αξιολόγηση του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου θα πρέπει να εδράζεται και στις αρχές και στις αξίες οι οποίες θα πρέπει να διέχουν τις πολιτικές μας και το διεθνές εμπόριο είναι μόνο μία πτυχή του των πολιτικών αυτών. Τώρα, έχουμε ένα τοπίο στο οποίο αλλάζουν συνεχώς οι προσδοκίες και θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε ε, να ε, το χρησιμοποιήσουμε καταλήλως αυτό. Η πρόκληση της χρήσης της οικονομικής ανάπτυξης για τους πολίτες μας είναι ουσιαστικός στόχος, ένας στόχος επί του οποίου το διεθνές εμπόριο και η οικονομική διπλωματία θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν και να βρούμε και κατάλληλους πόρους για αυτά. Επίση, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να εξετάσουμε με κριτικό βλέμμα κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει του πόρου ε, για να αντιμετωπίσει την αύξηση στι προσδοκίε για επικοινωνία για το εμπόριο. Πάντα αναφερόμαστε στην ανάγκη για διαφάνεια και ευπρόσδεκτη διαφάνεια, αλλά αυτό το οποίο ισχύει επίση είναι ότι ο κόσμο δεν περιμένει μόνο να του δίνονται πληροφορίε και να έχει πρόσβαση στι πληροφορίε με την κυριολεξία του όρου, αλλά να εισακούγεται κιόλα. Και νομίζω ότι ναι, μεν λογικό το αίτημα, αλλά αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις δομές που διαθέτει δεν είναι εξοπλισμένη για να την αντιμετωπίσει. Από τεχνική σκοπιάς ε, δεν ε, είναι απαραίτητα οι ίδιοι οι άνθρωποι που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα αιτήματα και μάλιστα ταυτόχρονα. Επομένως πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε πιο ευέλικτοι και θα πρέπει να διαθέτουμε τους πόρους για μια πιο σύγχρονη πολιτική εμπορίου στον 21ο αιώνα που βασίζεται σε αξίες και ε, ασχολείται με τους ενδιαφορομένους και να μην ξεχνάμε και τους πολίτες μας. Ευχαριστώ πολύ. Ο Χέλμουτ Σόλτς από πλευράς ΓΟΥΕ, όπως πάντα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή για την αναλυτική παρουσίαση της ε, πρότασης. Συμφωνώ με έναν άλλο στάνθο και εκείνον ότι πρέπει να σκεφτούμε πολύ σοβαρά ποια πρέπει να είναι η θέση μας ακριβώς για αυτή την προσπάθεια. Αφορά όχι μόνο την ε, Επιτροπή ε, Εξωτερικού Εμπορίου, αλλά όλους μας. Στο σημείο 4 ο εισηγητής αναφέρεται στις διάφορες περικοπές της κατηγορίας 4 και πρέπει να πούμε ότι ακόμη και στους τομείς όπου εμείς είμαστε υπεύθυνοι, στα μακροχρηματοδοτικά έχουμε πολλές ε, περικοπές. Θέλουμε να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη των χωρών που θέλουμε να υποστηρίξουμε. Και τι δίνουμε. Ε, δίνουμε με fast track χρήματα χωρίς να ελέγξουμε ποιες είναι οι προϋποθέσεις, ε, ποια είναι η κατάσταση στις χώρες θα επιτύχουμε να υπάρξει ε, βιώσιμη ανάπτυξη, θα επιτύχουμε να υπάρξει σταθερότητα σε αυτές τις κοινωνίες. Αυτό πρέπει να δούμε περισσότερο. Δεύτερον, κάτι άλλο που θέλουμε να προτείνουμε ως ομάδα, μέσω αυτής της πολιτικής μειώνονται τα τελωνιακά μας ε, έσοδα. Μπορεί τελικά να μην έχουμε καθόλου τελωνιακά έσοδα. Άρα πρέπει να δούμε από πού θα προκύψουν οι πιστώσεις που χρειάζεται η Ένωση για να προωθήσει κάποιες προσπάθειες προς το συμφέρον των πολιτών φυσικά. Υπάρχει αυτή η διαφορά. Πρέπει να καταστεί σαφής αυτή η διαφορά για όλους. ούτω ώστε να την κατανοήσει και ο ε, εισηγητής, οι εισηγητές που είναι αρμόδιοι στην Επιτροπή και προσβλέπω στη συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ισκά Κέλλερ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Συμφωνώ ότι το εμπόριο θα πρέπει να αποτελεί τμήμα της εξωτερικής μας πολιτικής ε, και να ε, μας ε, βοηθά να επιτύχουμε τους στόχους μας. Όμως, δεν είναι μόνο τα χρήματα, αλλά και οι πολιτικές τις οποίες ακολουθούμε. Και εμείς είμαστε υπεύθυνοι, οι πολιτικές αυτές, να συνάδουν με τους στόχου τη εξωτερική μα πολιτικής. Ασφαλώς, θα πρέπει να δούμε και την αξιολόγηση. Θα γίνεται μια διαρκής ε, αξιολόγηση για το τι βοηθάει την ανάπτυξη, για παράδειγμα, σε τρίτες χώρε και το κατά πόσον τα χρήματα που ξοδεύουμε βοηθούν προς αυτό. Σε ό,τι αφορά τα, τα κονδύλια έκτακτης ανάγκης, ε, συμφωνώ ότι το Κοινοβούλιο δεν θα πρέπει να είναι στο περιθώριο. Όμως θα πρέπει να σκεφτούμε πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε και την ευελιξία ταυτόχρονα. Γιατί καμιά φορά αυτά τα κονδύλια πρέπει να ε, δαπανώνται τάχιστα και χωρίς καθυστερήσεις. Θα κάνουμε κάποιες προτάσεις γι' αυτό. Δεν βλέπω να θέλει κανείς άλλο το λόγο, οπότε να δώσω το λόγο στην Κομισιόν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω και εγώ τον εισηγητή και τους ε, υπόλοιπους ε, ευρωβουλευτές ε, που παρενέβησαν και για την συνεχή τους στήριξη και όχι μόνο στον προπολογισμό. Αυτή τη στιγμή προετοιμάζουμε τις προτάσεις μας εμείς από πλευράς Κομισιόν. Η αναθεώρηση θα πρέπει να αποτελέσει ευκαιρία έτσι ώστε ο προπολογισμό να προσανατολιστεί προς την ανταγωνιστικότητα, ε, της, ε, την απασχόληση και την ανάπτυξη. Και βέβαια πολλά από όσα είπατε θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Θα δούμε τι ποσά θα έχουμε στη διάθεσή μας και πρέπει να αξιολογήσουμε το πώς, η ευελιξία του, πώς λειτουργεί η ευελιξία στο ισχύον πολιετές πλαίσιο και πώς μπορεί να βελτιωθεί. Τώρα, σε ορισμένα από τα πολύ συγκεκριμένα σημεία τα οποία θίξατε, για παράδειγμα, η συνεχής αξιολόγηση των διαφόρων πρωτοβουλειών. Είδα στο προσχέδιο έκθεσης ότι αναφέρεστε στην διεθνοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στη στήριξη προς τις επιχείρησεις γενικότερα. Συμφωνούμε μαζί σας. Θα πρέπει να αξιολογείται συνεχώς η προστιθέμενη αξία της χρηματοδότησης αυτής. Να σας υπενθυμίσω ότι οι Υπηρεσίε Κομισιόν μαζί με το Κοινοβούλιο σε τεχνικό επίπεδο συναντώνται τακτικά για να εξετάσουν τη χρηματοδότηση που δίδεται και αν αυτή έχει προσθέμενη αξία. Στον τομέα 4, εξωτερικές σχέσεις, που σας απασχολεί ιδιαίτερα, εκεί χρηματοδότηση σημαντικά περιορισμένη. Ε, αυτή τη στιγμή εκτιμούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ε, προκλήσεις και το πώς ε, θα αντιμετωπίσουμε το θέμα της ε, ενδιάμεσης αναθεώρησης. It was a Σύντομη απάντηση, κύριε Μπέγκε. Σας δίνω το λόγο. Yeah, thank you, Chair. I take note of the... Uh, Σημείωσα τη θέση της Κομισιόν. και θέλω να εκφράσω την ελπίδα μου ότι η Κομισιόν σε αυτές τις δυσχερείς διαπραγματεύσεις θα είναι στο πλευρό του Κοινοβουλίου και να μην τα παρατήσει ε, βεβιασμένα. Ξέρουμε όλοι ότι αυτές οι δυνατότητες ε, για, τους οποίους τόσο, για τις οποίες τόσο πολύ ε, πάλεψε το Κοινοβούλιο και οι οποίες μπόρεσαν να δημιουργηθούν μόνο μετά την ε, συμπληρωματική διαπραγμάτευση μέσω των τριών προέδρων, αυτή τη στιγμή έχουν πλήρως ε, εξαντληθεί. Δεν υπάρχει πλέον τίποτα διαθέσιμο. Δηλαδή η αξιοποίηση της ευελιξίας για να αντιμετωπιστούν οι ε, προκλήσεις που έχουμε ενώπιόν μας αποδεικνύουν ότι είχαμε δίκιο που ήμασταν επίμονοι για να υπάρξει περισσότερη ευελιξία αλλά έχει λήξει ήδη η χρηματοδότηση για αυτά τα νέα μέσα. Για το δεύτερο εξάμεινο δεν υπάρχει τίποτα πλέον. Για αυτά που είπε ο Σνάλφος Σόλτς τώρα. Για την κατάργηση των ε, ε, εσόδων από Βεβαίως ε, αυτό έχει επίπτωση στη συζήτηση για τη δομή των ιδίων πόρων. Και θέλουμε να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση. και υπάρχει μια κοινή έκθεση ΕΚΟΝ και, ε, και Μπούτζ για την ε, κοινή φορολογική ε, δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα το συζητήσουμε τώρα το θέμα αυτό, αλλά το θέμα πού θα βρούμε πόρους, ούτως ώστε στο μέλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, να έχει μέλλον και να έχει επαρκείς και σταθερούς πόρους. Αυτό το θέμα βέβαια θα μας απασχολήσει, αλλά σχετίζεται. Παρακαλώ την ε, Γραμματεία να παρακαλέσει την Επιτροπή να μας παρουσιάσει ένα κατάλογο των αποτιμήσεων και αξιολογήσεων που έχει κάνει το τελευταίο χρονικό διάστημα και τι προτίθεται να κάνει το επόμενο χρονικό διάστημα, τον επόμενο χρόνο, για να δούμε τι θα χρειαστούμε και για την ε, αναθεώρηση των πολιτών προοπτικών και για την ετήσια δημοσιονομική διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ. Θα το στηρίξουμε αυτό, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπέγκερ. Προθεσμία για τροπολογίες 25 Απριλίου, 12 το μεσημέρι. Και τώρα να δώσω το λόγο τον κύριο να δώσω συγγνώμη την Προεδρία στον κύριο Βίγκλερ για το σημείο 7. Τον Αντιπρόεδρο, κύριο Βίγκλερ. Uh, dear colleagues, so the next uh, item on the... Επόμενο σημείο της ημερησίας ε, διάταξης, ε, η εφαρμογή των συστάσεων του Κοινοβουλίου του 2010 σχετικά με τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εταιρική ευθύνη. Ο λόγος στην εισηγήτρια την κυρία Φορέντσα. ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τους ε, συναδέλφους ε, της Επιτροπής ε, καθώς και τους συναδέλφους των Επιτροπών που γνωμοδότησαν επί της έκθεσής μου. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τη Γραμματεία της Επιτροπής, τους κοιόδης ηγητές και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε ένα σημείο όπου ο πλούτος των τροπολογιών που υπευλήθησαν βοηθούν ε, τα όσα έχουμε λάβει από τους κοινωνικούς εταίρους και από τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Θεωρώ λοιπόν ότι είμαστε σε θέση να προωθήσουμε μία έκθεση που θα είναι στο ύψος των ε, περιστάσεων, ε, των προκλήσεων που προσπαθεί να αντιμετωπίσει η έκθεσή μας. Θα ήθελα εδώ να υποθυμίσω ένα στοιχείο για να ξεκινήσει η συζήτηση για αυτό το θέμα και να γίνει ανταλλαγή απόψεων. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε μία έκθεση η οποία στόχο έχει να εφαρμόσει τρεις προηγούμενες εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επομένω ε, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι περισσότερο υπεύθυνοι σε σχέση με τα όσα έχουν γίνει από το 2010 μέχρι σήμερα. Λαμβάνουμε φυσικά υπόψη μας και όλα, τα, όλα όσα έχουν συμβεί στο διάστημα αυτό. Πρόκειται για μια δύσκολη πρόκληση Προσπαθούμε να εφαρμόσουμε τρεις εκθέσεις και πρέπει να ε, έχει υπόψη του και το γεγονός ότι η εμπορική πολιτική είναι πάρα πολύ σημαντική για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για μια πιο βιώσιμη εμπορική πολιτική, αλλά και ε, στην εταιρική κοινωνική ευθύνη. Θα ήθελα λοιπόν σε αυτή την αντιαλλαγή απόψε να λάβουμε υπόψη κάποια κριτήρια τα οποία ε, είναι και αυτά τα οποία προσανατολίζουν το έργο μου. Καταρχάς, για ποιο λόγο γίνεται αυτή η έκθεση ίδια πρωτοβουλία. Πιστεύω ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη ε, τι εκκλήσει των μη κυβερνητικών οργανώσεων, ε, των συνδικάτων με τα οποία διαβουλευτήκαμε κατά τη σύνταξη αυτή τη έκθεση, να βλέπουμε μακριά. Να μην εξετάζουμε μόνο την βραχυπρόθεσμη εφαρμογή, που είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει, αλλά θα πρέπει το Κοινοβούλιο να σταθεί και στου στόχου τη έκθεση και σε διμερέ και σε πολυμερέ επίπεδο να αντιμετωπίσουμε ε, θεμελιώδη ζητήματα, όπως για παράδειγμα η μεταρρύθμιση των ε, ε, θεμάτων αυτών. Υπάρχουν ε, αρκετές τροπολογίες, να ευχαριστήσω τους συναδέλφους. Ε, δεν συμφωνώ με τις τροπολογίες οι οποίες περιορίζουν το επίπεδο της φιλοδοξίας μας. Θεωρώ όμως πολύ σημαντικές τις τροπολογίες οι οποίες στόχο έχουν να έχουμε πιο σημαντικά μέσα, να έχουμε συμβουλευτικές ομάδες για παράδειγμα ε, και να εφαρμόζονται οι ρήτρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τροπολογίες οι οποίες ε, αναφέρονται επίσης στη βιώσιμη ανάπτυξη. Εν να σας πω και το δεύτερο σημείο που με ενδιαφέρει. Πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να οπισθοδρομήσουμε σε σχέση με όσα έχουμε επιτύχει από πλευρά Κοινοβουλίου του 2010. Όλα όσα έχουμε επιτύχει πρέπει να ενισχυθούν, πρέπει να βελτιωθούν, αλλά να μην αποδυναμωθούν. Αναφέρομαι για παράδειγμα σε κάποιες τροπολογίες οι οποίες ε, θέλουν να είναι μικρότερη η δέσμευσή μας ε, στην ε, ε, κύρωση των 8 συν 4 συμβάσεων του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας. Επίσης, το να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στου κοινωνικού εταίρους. Αυτές είναι δεσμεύσει τις οποίες έχουμε αναλάβει και πρέπει να λογοδοτήσουμε για τα όσα έχουν συμβεί και όχι να περιορίσουμε την ε, έκταση και την εφαρμογή των μέσων αυτών. Ένα τελευταίο, το οποίο θεωρώ ότι είναι ουσιαστικό και αυτό, είναι να είναι πιο σημαντικός ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στις ε, εκτιμήσεις επιπτώσεων, αλλά και στην σύναψη εμπορικών συμφωνιών. Πιστεύω ότι η ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποτελεί πολύ σημαντικό άξονα των ε, εργασιών μας και κυρίως της έκθεσης αυτής. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι σαφής η πρόθεσή μου είναι μια φιλόδεξη έκθεση και είναι δύσκολο ε, στο χώρο που μας επιτρέπεται, τουλάχιστον στην πρώτη εκδοχή της έκθεσης, να συμπεριλάβουμε όλα αυτά τα τόσο σημαντικά σημεία ε, για την εφαρμογή τριών εκθέσεων. Ε, κλείνω με δύο πράγματα. Το πρώτο αφορά το GSP νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι για τρία στοιχεία. Πρέπει να δράσουμε πιο αποτελεσματικά στην παραβίαση των συμβάσεων στη βάση του συστήματος, επομένως να υπάρχει συμμετοχή ε, από πλευρά Κοινοβουλίου και να υπάρχει παρακολούθηση και να παρακολουθούν και κοινωνικοί εταίροι. Το δεύτερο μα ενδιαφέρει η ε, κοινωνική ευθύνη. Να ευχαριστήσω και τη Σκά Κέλλερ για τη βοήθειά τη. Δεν μπορώ να δεχτώ, ε, νομίζω, τροπολογίε οι οποίε μειώνουν τη δέσμευση του Κοινοβουλίου για τα θέματα αυτά. Πιστεύουμε ότι η δυνατότητα να υποστηρίξουμε κατάλληλες ενεργειακές πηγές είναι πάρα πολύ σημαντική για να επιτύχουμε και το στόχο που έχουμε ε, αναλάβει στο G20, δηλαδή τη μείωση της χρήσης των ορυκτών καυσίμων και πρέπει να υπάρχει συνονόηση από αυτόν. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τη συνάδελφο κ. Τόρνταρλινγκ για την πολύ σημαντική συνεισφορά της, ε, κυρίως ε, στο θέμα του CSR. Νομίζω ότι πρέπει να ξεχάσουμε την παροχημένη εφαρμογή του CSR, θα πρέπει να εφαρμοστεί με διαφορετικό τρόπο, για αυτή τη στιγμή έχουμε απλώς κάποιες εθελοντικές προσπάθειες προαιρετικά και δεν είναι και τόσο αποτελεσματικές για την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Από αυτή την άποψη νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνουν πολύ σημαντικά πράγματα και για την εταιρική κοινωνική ευθύνη η δέσμευσή μου ως εισηγήτρια, την οποία θα ήθελα να επαναλάβω εδώ για να ολοκληρώσω και την εισαγωγική μου παρέμβαση, είναι ότι είμαι απόλυτα διατεθειμένη να συζητήσω και με τους κοιόδης και με τους συναδέλφους. Θεωρώ ότι πρόκειται για μια πολύ σημαντική έκθεση, όχι μόνο για την εισηγήτρια και την, ε, ευρωπα και την Επιτροπή μας, αλλά και για όλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι η εμπορική πολιτική γίνεται σιγά σιγά ένα όλο ένα και πιο σημαντικό κεφάλαιο της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Uh, thank you very much, Ευχαριστώ πολύ. Πληροφοριακά να σας πω ότι 219 τροπολογίες έχουν κατατεθεί, το είπε και η συγγήτρια, και περίπου 100 ακόμα από τις νομοδοτούς επιτροπές. Τέσσερις επιτροπές. Ε, ΑΦΕΤ, και ΕΜΠΛ. Ο κ. Φίσας εκ μέρους του ΕΛ καταρχήν. Ευχαριστώ. Κ. Σαϊφή, ε, λυπάται για την απουσία της. Βρίσκεται σε επίσημη αποστολή στο εξωτερικό, οπότε μου ζήτησε να πάρω εγώ το λόγο εκ μέρους της. Ο στόχος της έκθεσης είναι να υπογραμμίσει τις ε, δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 2010 ε, προκειμένου να κάνει μια, και ένα απολογισμό υπογραμμίζοντας τους ε, στόχους και τις δράσεις που θα πρέπει να ακολουθούν. Σε, σε σχέση με τις τροπολογίες κυρία Σαϊφή, πρόκειται για τροπολογίες που έχουν ως στόχο να υπενθυμίσουν ότι το εμπόριο επιτρέπει να προωθήσουμε και να προστατεύσουμε τις αρχές, ε, τις αξίες συγγνώμη, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στη διεθνή σκηνή και να εξασφαλίσουμε την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προδιαγραφών. Από αυτή την έννοια η ύπαρξη ε, κεφαλαίου για την βιώσιμη ανάπτυξη στις εμπορικές συμφωνίες είναι μεγάλη σημασία και θα πρέπει να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε μια συνεργασία σε πολυμερές επίπεδο για αυτό το θέμα μαζί με άλλους διεθνείς παίκτες ε, όπως ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας, ε, το ΩΣΑ κλπ. Σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να μεριμνήσουμε έτσι ώστε ρήτρε ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είναι παρούσε ε, σε διεθνεί εμπορικέ συμφωνίε να ε, τυχάνουν σεβασμού και να εφαρμόζονται. Γι' αυτό το λόγο είναι σημαντικό να παρακολουθούμε στενά και σε βάθο ε, την εφαρμογή αυτών των ρητρών. Αυτό εμπλέκει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την κοινωνία των πολιτών. Υπ' αυτή την έννοια έχουμε επαναλάβει το αίτημά μας ε, να διοργανωθούν φόρα για την βιώσιμη ανάπτυξη ή συμβουλευτικές ομάδες ε, προκειμένου να διαπιστώνουμε το αν οι διεθνείς συμφωνίες ε, τηρούνται και σε επίπεδο ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σε επίπεδο κοινωνικών και περιβαλλοντικών προδιαγραφών. Προτείνουμε συγκεκριμένες δράσεις, τις οποίες θα υλοποιούμε σε συνεργασία με τους εταίρους μας ε, για να διορθώσουμε ε, αστοχίες στην εφαρμογή αυτών των εμπορικών συμφωνιών. Επίσης, ζητούμε να γίνει αναφορά στο σύστημα των γενικευμένων προτιμήσεων ΣΥΝ. Αυτό το σύστημα βοηθάει στην ε, προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του, περιβάλλοντος. Ε, η καταπολάμηση της καταναγκαστικής εργασίας και της εργασίας των παιδιών ε, είναι θέματα τα οποία θα θέλαμε να υπογραμμιστούν στην έκθεση. Ζητούμε από την Κομισιόν να αναλάβει δράση και προτείνουμε στις εμπορικές συμφωνίες να συμπεριλάβουμε και το στόχο και τους δύο αυτούς ε, στόχους εντάσσοντάς τους στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω μιας ε, νομοθετικής ε, πρότασης ισορροπημένης και ρεαλιστικής όπως είχαμε ζητήσει το 2010. Επίσης, έχουμε υποβάλει τροπολογίες σε ό,τι αφορά την εταιρική κοινωνική ευθύνη προκειμένου να υπενθυμίσουμε την, ε, το σύμφωνο Ε, το, το ε, πρόγραμμα της Γκράνα Πλάθα του Πακιστάν και να το διευρύνουμε και σε άλλες περιοχές. Ε, η, ε, επίσης οι πρωτοπολογίες μας αφορούν γενικότερα τη στρατηγική μας ό,τι αφορά την κοινωνική ευθύνη. Ευχαριστώ. Η Κρήτον Ντάλινγκ για τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ και τον εισηγητή το γεγονό ότι υπήρξαν τόσε τροπολογίε αποδεικνύουν ότι οι συνάδελφοι θεωρούν ότι είναι σημαντικό το θέμα για μα, του σοσιαλιστέ. Είναι βασικό πυλώνα μια ε, δίκαιη εμπορική πολιτική. Ελπίζω ότι οι διαπραγματεύσει για ένα συμβαστικό κείμενο θα ε, ικανοποιήσουν και αυτούς που δεν είναι εδώ, που περιμένουν ακριβώς να γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματά τους στις εμπορικές συμφωνίες. Για ορισμένους είναι θέμα ζωής και θανάτου και υγείας. Είναι σημαντική έκθεση, πρέπει να αντιμετωπιστεί με υπεύθυνο τρόπο. Μαζί με τους συναδέλφους μου από την ομάδα μου υπέβαλα δύο ομάδες τροπολογιών, μία για να υπάρξει μια εξισορρόπηση της έκθεσης, ούτως ώστε να κάνει αξιολόγηση του τι επέτυχε και πού απέτυχε η Κομισιόν για να ανταποκριθεί στα αιτήματά μας από το 2010. Και η άλλη ομάδα προτείνει νέες ιδέες μετά τα πρώτα χρόνια εφαρμογής ε, των ε, συμφωνιών αυτών με τα κεφάλαια για την βιώσιμη ανάπτυξη και ε, εκφράζει νέες ανησυχίες που προέκυψαν από πρόσφατες εξελίξεις. Για παράδειγμα τα τραγικά γεγονότα στο Ράνα Πλάζα και επίσης τις προτάσεις του ΟΣΑ για τις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας. Υπάρχουν πολλές προτάσεις από καλές από μερικές ομάδες, αλλά άλλες θα μας επανέφεραν στην κατάσταση πριν από το 2010. Η αξιοπιστία μας ε, θα ετίθετο σοβαρά εν κινδύνο, αν αυτοϋπονομευθούμε. Η διαδικασία επίτευξης συμβαστικών τροπολογιών μόλις έχει ξεκινήσει, ελπίζω να είναι επικοδομητική. Η έκθεση αυτή έχει καθυστερήσει πάρα πολύ. Οποιαδήποτε περαιτέρω μείωση της σημασίας των αναφορών στην εταιρική κοινωνική ευθύνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα στις εμπορικές συμφωνίες θα ήταν απαράδεκτη. Η κυρία Μάλστρομ έχει πει ότι τα θέματα αυτά είναι προσωπική της προτεραιότητα. Πρέπει να αξιοποιήσουμε την έκθεση αυτή για να πούμε συγκεκριμένα τι αναμένουμε και από εκείνη και από την Επιτροπή γενικότερα και γιατί θεωρούμε ότι οι προτεραιότητες αυτές πρέπει να είναι αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης με τη συμμετοχή των αφορομένων ούτω ώστε τα λόγια μα να γίνουν πραγματικά πράξη. ECR, e uh, e εδώ ο αντιπρόεδρος μας κύριος Ζαχράντιλ. Ευχαριστώ πρόεδρε συνάδελφοι. Έχουμε μια μακροχρόνια προσέγγιση υπέρ του εμπορίου, υπέρ των επενδύσεων. Έτσι θεωρώ ότι επιτυχάνουμε πολύ περισσότερα και για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για τα κοινωνικά δικαιώματα και για τα περιβαλλοντικά ε, στάνταρ γιατί θεωρούμε ότι οι αντισυμβαλόμενοι είναι ισότιμοι εταίροι. Τους επιτρέπουμε λοιπόν να δεσμευτούν οι ίδιοι ότι θα βελτιώσουν την κατάσταση σε αυτούς τους τομείς παράλληλα αναπτύσσοντας την πολιτική τους για το εμπόριο και τις επενδύσεις. Για να είμαι λοιπόν ε, ειλικρινής. Δεν μας ικανοποιούν ε, ορισμένες τροπολογίες αλλά και ορισμένες τάσεις της αρχικής έκθεσης που θα μπορούσα να τη χαρακτηρίσω πολιτικοποίηση του εμπορίου. Μπορώ να υποστηρίξω την εισηγήτρια όταν τονίζει ότι πρέπει να παρακολουθούμε και να βλέπουμε πώς εφαρμόζονται οι συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου. Αλλά αυτή η πολιτικοποίηση του εμπορίου θεωρούμε ότι είναι αντίθετη προς τους στόχους μας, ε, αναποτελεσματική και ενδεχομένως ζημιογόνος. Ε, ιδιαίτερα δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με τον συνδυασμό των μελλοντικών συμφωνιών εμπορίου με δεσμευτικές αποτιμήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν καταλαβαίνω το γεγονό ότι δεν καταλαβαίνω πώς θα λειτουργούσε ένας μηχανισμός επίλυσης ε, διαφορών που θα ήταν άμεσα προσβάσιμος στους κοινωνικούς εταίρους. Πρέπει να διευκρινιστούν αυτά τα πράγματα. Επίσης για τις κυρώσεις και αναστολές ε, των συμφωνιών που προτείνονται, ανάλογα με τις ε, περιστάσεις, έχουμε επιφυλάξεις. Και ως συνήθως, είμαστε συστηματικά αντίθετοι προς την δεσμευτική προσέγγιση που προτείνεται για την κοινωνική εταιρική ευθύνη και έχουμε υποβάλει τροπολογίες προς αυτή την κατεύθυνση. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές απόψεων. Αλλά παρόλα αυτά θέλουμε να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις, θέλουμε να συμμετάσχουμε στις διαπραγματεύσεις, θέλουμε να επιτύχουμε συμβιβασμούς, τουλάχιστον στους τομείς που αφορούν την αποτελεσματική εφαρμογή των υπαρχουσών συμφωνιών, μηχανισμούς ε, GSP-SYN, Και μπορώ να πω ότι θέλουμε να γίνει η επόμενη συνάντηση των σκιωδών όπου θα συμβάλλουμε επικοδομητικά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. Φιλελεύθερη. Χάνου Τάκουλα. Ε, ε, μιλώ εκ μέρους της κυρίας Δεσάρν πάνω από 200 τροπολογίες υποβλήθηκαν ε, και εμείς συνεργαζόμαστε για 20 περίπου, πάνω από 20 ε, συμβαστικές τροπολογίες. Επιθυμούμε το ψήφισμα να βασιστεί στις συστάσεις του Κοινοβουλίου του 2010. Και θα θέλαμε μάλιστα στο θέμα της εταιρικής συνολικής ευθύνης να είμαστε ακόμα πιο φιλόδοξοι. Τα βασικά σημεία τα οποία θα πρέπει να μπουν στο τελικό κείμενο είναι τα εξής. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παίξει ένα δραστήριο ρόλο στην υιοθέτηση, στην υλοποίηση των στόχων ε, ε, ε ανάπτυξη 2030 του ΟΗΕ. Δεύτερον, τα θέματα των γυναικών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην καινούργια εμπορική στρατηγική της Ευρωκομισιόν. Θα πρέπει να γίνεται συστηματική αξιολόγηση αντικτύπου ε, πριν από οποιαδήποτε εμπορική διαπραγμάτευση. Θα πρέπει να εξετάζονται τα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και να δίδεται ιδιαίτερη σημασία πιο ευάλω, στα πιο ευάλωτα τμήματα του πληθυσμού. Είτε είναι μειονότητες, ε, είτε ε, επειδή ε, για κάποιο λόγο φύστανται διακρίσεις. ιδιαίτερα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι πιο απομακρυσμένες περιοχές, και να γίνεται μια αξιολόγηση που δεν γίνεται τακτικά αυτή τη στιγμή. Η εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να συνεισφέρει στην ενεργειακή μετάβαση. Στην, ε, η πρωτοβουλία για τα πράσινα αγαθά, για παράδειγμα, είναι ένα σωστό βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση. Τέλος, θα πρέπει επίσης να ε, ε, να ενισχυθούν συνεργασίες όπως ε, ε, πρωτοβουλίες όπως η, η, η, η οικολογική σήμανση, ε, η υποχρεωτική κοινοποίηση πληροφοριών έτσι ώστε οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να είναι πιο υπεύθυνες οικολογικά και κοινωνικά. Uh, thank you very much. And, uh, for the Greens... Για τους πράσινους Ισκάκελερ. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ την εισηγήτρια για την εξαιρετική της έκθεση. Έχουμε υποβάλει κάποιες τροπολογίες και από πλευράς μας ε, θα πρέπει σίγουρα να εφαρμόζεται η ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εάν έχουμε συμφωνία για όλα τα υπόλοιπα, τότε τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να εφαρμόζονται, πρέπει να επιβάλλονται κυρώσει, και αν θέλουμε να εφαρμόσουμε και τη νέα στρατηγική για μεγαλύτερη έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα, πρέπει να εφαρμόζονται και αυτά και η εταιρική κοινωνική ευθύνη. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά για μας. Τώρα, για αυτά τα οποία έχει ήδη συστήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να υπάρχει ε, απαγόρευση των εισαγωγών όταν υπάρχει καταναγκαστική εργασία. Αυτό είναι κάτι το οποίο ισχύει εδώ και καιρό, αλλά μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει κάνει κάτι για την εφαρμογή του. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι είναι ευκαιρία να το συμπεριλάβουμε και αυτό στην έκθεση και ε, θα θέλαμε και απάντηση από αυτού όσον αφορά το περιβάλλον και το εμπόριο. Υπάρχουν τροπολογίε για να γίνει έκκληση κυρίω προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σταματήσει να ασχολείται με ε, εμπορικές συμφωνίες ε, για να μπορέσει να εξυπηρετήσει η πολιτική εμπορίου του στόχους της κλιματικής αλλαγής και όχι να τους υποσκάπτει. Επίσης, ε, έχει γίνει κάποια πρόοδος ε, για τη διάκριση μεταξύ των προϊόντων τα οποία χρησιμοποιούνται και τις μεθόδους παραγωγής δεν έχουμε δει καμία πρόοδο τα τελευταία 6 χρόνια. Ίσως λοιπόν και αυτό θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη. Το Κοινοβούλιο στο παρελθόν είχε ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο προσαρμογής ε, των δασμών. Ε, και πάλι ζητήθηκε να ε, εκμεταλλευτούμε το μέσο αυτό στην ε, μεταρρύθμιση του συστήματος εμπορίας εκπομπών. Ίσως θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε και εδώ, ώστε επιτέλους να υλοποιηθεί. Επίση, ζητάμε να συμπεριλάβουμε στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία οδηγίες ε, του ΟΣΑ και των ε, Ηνωμένων Εθνών για τις ε, αλυσίδες διανομής, για το πώς τις λαμβάνουμε υπόψη, πώς διασφαλίζουμε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και εταιρική κοινωνική ευθύνη γίνονται σεβαστά σε αυτό το επίπεδο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη στρατηγική και πρέπει να πούμε κάτι γι' αυτό και στην έκθεσή μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Η Τιτσιάνα Μπεγκίν από το EFTD. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ την εισηγήτρια για τα όσα έχει κάνει. Και θα ήθελα να συνοψίσω λίγο τη συζήτηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπου συνέταξα τη γνωμοδότηση για την έκθεση αυτή. Και εγώ και άλλες πολιτικές ομάδες θεωρήσαμε ότι είναι απαραίτητο να ξεκινήσουμε από ένα σημείο που για μας είναι υψίστης σημασίας. Να σέβεται η εμπορική μας εταίρη του 8 βασικούς κανόνες για την εργασία και τις 4 ε, συμβάσεις που αποτελούν προτεραιότητα του Διεθνούς Οργανισμού Εργασία. Αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται στις συνθήκες μας και σε όλες τις ε, διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να υπάρχει μια κοινωνική ρήτρα που θα εγγυάται την εφαρμογή. Αλλά δεν φτάνει αυτή η ρήτρα. Εχθές παρενέμει στην Επιτροπή Απασχόλησης για να καταγγείλω τις ε, πρακτικές εργασίες ε, στη Νότια Κορέα και την, τι γίνεται με τους ακτιβιστές σε περιβαλλοντικό επίπεδο. Πρέπει να υπάρχει κατάλληλη αντιλογή με την Ευρώπη, η οποία υπόσχεται να σεβαστεί τα δικαιώματά τους και τελικά δεν υπάρχει κατάλληλη εφαρμογή. Το να υπάρχει ρήτρα είναι απαραίτητο, αλλά είναι άχρηστη η ρήτρα αυτή αν δεν παρακολουθεί τη εφαρμογή τη. Πρέπει να δούμε λοιπόν και τι γίνεται με τη βιώσιμη ανάπτυξη στι διμερεί και πολυμερεί συμφωνίε, να υπάρχει ένα μηχανισμό ελέγχου, ο οποίο θα είναι ανοιχτό και στου κοινωνικού εταίρου και να υπάρχουν και μηχανισμοί κυρώσεων εάν δεν εφαρμόζονται. Ένα άλλο σημείο για το οποίο είμαι περήφανη είναι το σημείο στο οποίο εμεί ζητάμε η ρήτρα αναστολή που υπάρχει στι διμερεί συμφωνίε να ενεργοποιείται όταν υπάρχουν πολύ σοβαρέ παραβιάσει των στόχων ή των ε, κοινωνικών και περιβαλλοντικών κανόνων, διότι επιτρέψτε μου να πω ότι δεν ε, χρησιμεύει σε τίποτα να κονίζουμε τα δόντια μας εάν δεν μπορούμε στη συνέχεια να δαγκώσουμε. Και εγώ και οι συνάδελφοι στην Επιτροπή Επασχάλησης θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχουν κίνητρα για να δώσουμε ε, τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να εφαρμόζουν κοινωνική εταιρική ευθύνη ε, για να είναι οι πρώτες οι οποίες ε, θα εφαρμόζουν μέτρα όταν υπάρχουν προβλήματα σε περιβαλλοντικό και κοινωνικό επίπεδο και στις θηγατρικές τους εταιρείες. Επίσης, ε, προσπαθούμε να έχουμε κάτι αντίστοιχο με αυτό που έχουμε για τα ε, ορυκτά σε περιοχές σύγκρουσης και να υπάρχει και κατάλληλο προσωπικό για να μπορούμε να κάνουμε επιθεωρήσεις εργασίες. Ορισμένα από αυτά τα πράγματα υπάρχουν στο κείμενο της εισηγήτριας και εγώ ελπίζω ότι οι αρχές της γνωμοδότησής μας, οι οποίες ε, εγκρίθηκαν με ευρία πλειοψηφία, θα γίνουν δεκτές από την εισηγήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Ωραία. Από τους συναδέλφους υπάρχει κάποιος κάτι που θα ήθελε κάτι να προσθέσει. Αν όχι, να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να κάνει κάποιες σύντομες παρατηρήσεις. Από τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου είναι εδώ η Σίλβια Φορμεντίνη. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για όλα σας τα ενδιαφέροντα σχόλια που κάνατε. Θα είμαι σύντομη. Πρώτον να υπενθυμίσω ότι η Κομισιόν ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τις εργασίες του Κοινοβουλίου για αυτό το θέμα. Ε, είναι, προτεραιότητα για μας, τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η εταιρική κοινωνική ευθύνη. Να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και τους άλλους ε, ε συναδέλφους που είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν με την Κομισιόν. Θα είναι πολύ χρήσιμο αυτό. Οι σημερινές συζητήσεις και ο μεγάλος αριθμός ε, τροπολογιών που έχουν υποβληθεί ε, επιβεβαιώνουν τον ε, πλούτο και τη σημασία του θέματος. Αλλά το θέμα είναι επίσης και πολύ περίπλοκο. Δεν θέλω να μπω σε λεπτόμερη σχόλια για κάθε τροπολογία προφανώς, αλλά να κάνω κάποια βασικά σχόλια. Πρώτον, η Κομισιόν καλωσορίζει το γεγονό ότι πολλέ τροπολογίε προτείνουν να αναγνωριστούν όσα έχουν επιτευχθεί στο παρελθόν παράδειγμα η υπεύθυνη εταιρική συμπεριφορά ε, κλπ. Επίσης ε, κάποιες τροπολογίες καλύπτουν νέες εξέλιξεις ε, που δεν είχαν καλυφθεί παλιότερα. Για παράδειγμα το σύμφωνο του Μπαγκλαντές. Επίσης καλωσορίζουμε το γεγονός ότι πολλές τροπολογίες υπογραμμίζουν το έργο σε συνεργασία με διεθνή όργανα και φορεί. Θα πρέπει να συνεχίσουμε προ αυτήν την κατεύθυνση. Επίση, καλωσορίζουμε το γεγονό ότι ορισμένε τροπολογίε προσπαθούν να εξισορροπήσουν ε, αυτό που μπορεί να κάνει και έχει κάνει η, πολιτική, η εμπορική πολιτική και αυτό μπορούν να κάνουν ή έχουν κάνει άλλε πολιτικέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, για παράδειγμα, η αναπτυξιακή πολιτική. Ορισμένε τροπολογίε ε, έχουν κάποιε ανακρίβειες ε, ε, στα στοιχεία τα οποία παρουσιάζουν. Ελπίζω ότι αυτό θα διορθωθεί στις διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν. Αυτά, μια και δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Ένα τελικό σχόλιο. Επαναλαμβάνω ότι είμαστε διαθέσιμοι και ενδιαφερόμαστε να συνεχίσουμε το διάλογο όπως νομίζετε πιο κατάλληλο. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πολύ σύντομα, επειδή δεν, δεν έχουμε τόσο πολύ χρόνο, ε, να επανέλθω στην εισηγητριά μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που έλαβαν το λόγο, τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου και τη Γραμματεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπ... της Επιτροπής μας. Δύο διευκρινήσεις ε, για τη μέθοδο εργασίας επαναλαμβάνω αυτό που σας έλεγα, για μένα είναι πολύ σημαντικό στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης των τροπολογιών, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει, θέλω να συμμετέχουν όλοι και όλες, διότι θεωρούμε ότι επειδή είναι τόσο σημαντικό το θέμα αυτό, θα πρέπει να βρούμε μία λύση με τη μέγιστη δυνατή συνένεση. Το δεύτερο θέμα αφορά τα χρονοδιαγράμματα. Εδώ υπενθυμίστηκε πόσες ε, πολλές ε, και ποιοτικέ είναι οι τροπολογίες που υπευλήθησαν και πόσο σημαντικό είναι το ζήτημα το οποίο ε, εξετάζουμε σε αυτές τις τρεις εκθέσεις τις οποίες ενοποιούμε σε μία έκθεση Γι' αυτό άλλωστε και δεχτήκαμε την πρόκληση. Αντί να ψηφίσουμε απευθεία σήμερα, προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτό το επιπλέον βήμα, το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, μια ανταλλαγή απόψεων για τις τροπολογίες δηλαδή, για να μπορέσουμε να μας δώσουν και τις γνωμοδοτήσεις τους οι άλλες επιτροπές. Τελευταία η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, η οποία μας την έστειλε τη Δευτέρα. Επομένως υπήρχε μια παράταση ε, που δεν ήταν ευθύνη ουσιαστικά κανενός, αλλά ήταν λόγω της σημασίας των θεμάτων που εξετάζουμε. Για να συνοψίσω σε αυτά που είπαν οι συνάδελφοι, και εγώ Πιστεύω ακράδαντα ότι το θέμα της βιώσιμης ανάπτυξης ε, θα πρέπει να αποτελεί το κεντρικό θέμα στην ε, έκθεση, όπως επίσης άλλωστε αναφερόταν στην έκθεση και το θέμα της καταπολέμησης της ε, εργασίας των ανηλίκων. Όσον αφορά αυτό που έλεγε συνάδελφος Κίρτολ Ντάρλινγκ, και εγώ πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει κατάλληλη ισορροπία και να ε, ζητήσουμε να τηρηθούν όλα όσοι έχει κάνει η Επιτροπή από το 2010 μέχρι σήμερα. Συμφωνεί και εκπρόσωπο τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου. Θα πρέπει να επισημάνουμε και τα θετικά στοιχεία, όπω για παράδειγμα ε, το σύμφωνο για το Μπαγκλαντέ. Και θεωρώ επίσης ότι πρέπει ε, όταν θα συζητήσουμε τις τροπολογίες να δεχτούμε και όλες τις νέες προτάσεις για το βιώσιμο εμπόριο θεωρώ ότι έτσι και πραγματικά τελειώνω με αυτό, θα μπορέσουμε να έχουμε μία συγκεκριμένη ε, πρόταση μέσα αυτής της έκθεσης. Και εδώ ε, συμφωνώ με το πνεύμα της παρέμβασης της συναδέλφου Μπεγκίν. Ε, σημαίνει ότι πρέπει το Κοινοβούλιο να έχει αποτελεσματικά μέσα που δεν σημαίνει, για να απαντήσω και στο συνέδελφο, ότι πολιτικοποιούμε το εμπόριο. Σημαίνει απλώς ότι αποφασίζουμε αν θέλουμε να έχουμε ε, κάποια μέσα τα οποία θα είναι δεσμευτικά για τις ε, ρήτρε των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, και για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ευχαριστώ την ε, συνάδελφο Κέλλερ και για την πρότασή της για το θέμα της δουλείας και το πώς μπορούν να εφαρμόζονται οι ρήτρε για τα ανθρώπινα δικαιώματα και επίσης να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τη συνάδελφο Μπεγκίν και τα όσα έχει κάνει ε, όλη η Επιτροπή, διότι το θέμα των συμβάσεων ε, του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας και της ρήτρα ανιστολής είναι πάρα πολύ σημαντικό ώστε να αποφύγουμε η έκθεση αυτή και εν γέννη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει μια στάση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη βιώσιμη ανάπτυξη η οποία θα είναι πολύ προηγμένη σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά στην πράξη θα είναι λίγο αποτελεσματική. Εμείς θέλουμε το αντίθετο. Θέλουμε να υπάρχει αντιστοιχία ανάμεσα στην ε, βούληση να έχουμε ε, ε, μια εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία θα λαμβάνει υπόψη της και τα ανθρώπινα δικαιώματα και να είναι αυτό κάτι το οποίο θα βοηθάει και τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής. Ευχαριστώ. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας θα γίνει στις 23 και 24, στη συνεδρίαση 23-24 Μαΐου και θα δούμε πότε θα γίνει η ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Ε, έκλεισε αυτό το θέμα. Να περάσω στο επόμενο θέμα. Με συγχωρείτε αγαπητοί συνάδελφοι, δεν τα πάω τόσο καλά ως πρόεδρος της ΙΝΤΑ, γιατί δεν τηρώ τα προβλεπόμενα χρονικά όρια. Πρέπει λοιπόν ε, να αξιοποιήσουμε καλύτερα το χρόνο που μας μένει. Έχουμε τώρα μια νέα μακρόπνη και, και μελλοντική στρατηγική για το εμπόριο και τις επενδύσεις. Όπως ξέρετε, βασίζεται στην ανακοίνωση που παρουσίασε στην Επιτροπή μας η Επίτροπος ε, ε, Μάλστρομ, εμπόριο για όλους, τον περασμένο Οκτώβριο για το μέλλον της στρατηγικής για το εμπόριο και τις επενδύσεις αποφασίσαμε να συντάξουμε μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλία. Τη συζητήσαμε στη συνεδρίασή μας το Φεβρουάριο και τώρα στρέφομαι προς την εισηγήτρια τη συνάδελφο Τιτσιάνα Μπέγκη να παρουσιάσει το σχέδιο έκθεσης. Παρακαλώ Τιτσιάνα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Επιτροπή για το έγγραφο το οποίο αναφέρατε, το οποίο είναι και ενδιαφέρον και απαραίτητο. Και να ευχαριστήσω και εσάς κύριε Πρόεδρε, τους συναδέλφους συντονιστές και τους ε, σκιώδης ηγητές που μου εμπιστεύτηκαν το θέμα αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση περίμενε εναγωνίω αυτό το στρατηγικό και προγραμματικό έγγραφο. Για λόγους χρόνους δεν θα σταθώ πολύ στι αρκετές πτυχές ε, του εγγράφου της Επιτροπής που θεωρώ ότι είναι σημαντικά, αλλά θα σταθώ σε αυτά τα οποία θέλησα να συνεισφέρω εγώ. Ο τίτλο είναι πολύ αντιπροσωπευτικό εμπόριο για όλους, προς μια πιο υπεύθυνη εμπορική πολιτική. Η ευθύνη είναι μια υπέροχη λέξη με πολλές ερμηνείες, αλλά για να μην μείνει κενό γράμμα θα ήθελα να αναφερθώ στον όρο αυτό. Ευθύνη σημαίνει λογοδοτό. Λογοδοτό στον ελεγκτή που είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά οι ίστατοι ελεγκτέ είναι οι πολίτες οι οποίοι πρέπει να ελέγχουν, ε, αλλά πρέπει να γνωρίζουν για να ελέγχουν. Γι' αυτό ακριβώ και η ευθύνη είναι, ε, συμβαδίζει με τη διαφάνεια που πρέπει να εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα. Η πρωτοβουλία τη διαφάνεια που έχει ήδη αναλάβει η Επιτροπή πρέπει να χρησιμοποιούνται σε όλε τι εμπορικέ συμφωνίε συστηματικά. Η συνεργασία με το Κοινοβούλιο και του πολίτε πρέπει να είναι συνεχής και μόνιμο. Το Συμβούλιο πρέπει επίση να συνεχίσει τι καλέ πρακτικέ τη ε, δημοσίευση των ε, διαπραγματευτικών εντολών, διότι μόνο ο ενήμερο ελεγκτής είναι ο αποτελεσματικός ελεγκτής. Ευθύνη σημαίνει να αναγνωρίζω το ρόλο μου στο εσωτερικό ενό περιφερειακού και παγκόσμιου συστήματο πολύ περίπλοκου και να δρούμε αναλόγω. Η εμπορική πολιτική εγγράφεται σε ένα πιο μεγάλο και περίπλοκο σύστημα και πρέπει να συνάδει και με τι άλλε εξωτερικέ πολιτικέ. Οι εμπορικέ επιλογέ έχουν πολύ βαθιές συνέπειε και είναι ουσιώδεις για να αντιμετωπίσουμε τη μετανάστευση. Χάρη στη δύναμή τη, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μεγάλη βαρύτητα στι ε, παγκόσμιες αλυσίδε τη αξία και επομένω πρέπει να χρησιμοποιήσει αυτή τη βαρύτητα για να προωθεί τι δικέ τη αξίε, χωρί να χάσει καμία ευκαιρία για να το υλοποιήσει αυτό. Οι συνάδελφοι που αναφέρθηκαν σε διαπραγμάτευση για τα ορυκτά σε περιοχέ σύγκρουση είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Ε, ευθύνη σημαίνει να κάνω και το καθήκον μου, ακόμα και όταν είναι δύσκολο, διότι η εμπορική πολιτική πρέπει να κάνει περισσότερο για να προεθήσει το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κοινωνικού και περιβαλλοντικού κανόνε και την εταιρική κοινωνική ευθύνη και ένα ε, παγκόσμιο σύστημα το οποίο θα βασίζεται στο σεβασμό των κανόνων. Ελπίζω λοιπόν ότι όλε οι συμφωνίε ελευθέρων συναλλαγών έχουν κεφάλαια για την βιώσιμη ανάπτυξη, τα οποία είναι δεσμευτικά και αποτελεσματικά και πλευλέπουν και ρήτρε ε, ε, αναστολής και μηχανισμούς μέσω των οποίων μπορούμε να ζητήσουμε επισήμως εμείς οι ε, και οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών έρευνες για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η εμπορική πολιτική πρέπει να περιλαμβάνει και τους πιο δυνάμους. 780 εκατομμύρια ανθρώπων που ζουν κάτω από το επίπεδο της φτώχειας. 865 εκατομμύρια γυναίκες που δεν συμμετέχουν στην οικονομική ζωή των χωρών τους και γι' αυτό η στρατηγική θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της και την ένδια και τα θέματα φύλου. Ευθύνη επίσης σημαίνει σεβασμό σεβασμό. Σεβασμό της διάθεση των πολιτών και αυτών που την εκφράζουν. Γι' αυτό και ζητώ ε, το κείμενο αυτό να έχει μια ενισχυμένη εταιρική σχέση μεταξύ Επιτροπής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό δεν σημαίνει μόνο ότι πρέπει να ενημερώνεται το Κοινοβούλιο, αλλά θα πρέπει να συμμετέχει ε, σε όλα τα στάδια τη εμπορική πολιτική πέραν των ε, νόμιμων υποχρεώσεων που αναγράφονται στι συνθήκε. Να σέβονται τι θέσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σημαίνει ότι θα πρέπει να σέβονται τη βούληση των Ευρωπαίων πολιτών. Τα ψηφίσματα για τις ε, συμφωνίε, ε, οι οποίες είναι υποδιαπραγμάτευση σημαίνει ότι σεβόμαστε την Ευρωπαϊκή Κοινογνώμη και λεπόμαστε που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ε, λαμβάνει υπόψη τις, τις συμφωνίες. Όπως για παράδειγμα τη συνέχεια του ψηφίσματος για την ΤΙΣΑ όπου λέει ότι δεν θέλει να δώσει συνέχεια στο αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να υπάρχει ένας θετικός κατάλογος και για την πρόσβαση στην αγορά και την εθνική αντιμετώπιση. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει ένα σαφές αίτημα. Η Ευρώπη δεν πρέπει να εφαρμόζει τη προσωρινά πριν να τα έχει εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η ευθύνη είναι και ευθύνη προς τους εμπορικούς μας εταίρους, η οποία εκφράζεται στην αναγνώριση του πολυμερού συστήματος ως την καλύτερη επιλογή για να εγγυηθούμε ανοιχτό, νόμιμο και θεμητό εμπόριο που θα βασίζεται στους κανόνες και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει μια στοχευμένη περιφερειακή στρατηγική, κυρίως όσον αφορά την Ασία και τη Λατινική Αμερική αλλά η ευθύνη είναι και προ του Ευρωπαίου πελίτε, οι οποίοι θα πρέπει να προστατεύονται από του κινδύνου αυτών οι οποίοι δεν ε, σέβονται του κανόνε και απειλούν τον τρόπο ζωή του. Γι' αυτό ακριβώ πρέπει να είμαστε στεναροί στο αίτημα μεταρρύθμιση του συστήματο τη εμπορική προστασία και να είμαστε ε, κατάφορα αντίθετοι στην, ε, στο καθεστώ οικονομία τη αγορά στην Κίνα. Ε, αλλά οι πολίτε μα πρέπει να υποφελούνται και από τα πολύ μεγάλα πλεονεκτήματα που μπορεί να του προσφέρει το εμπόριο. Μόνο το 13% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ε, δραστηριοποιείται εκτό των συνόρων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ε, ο αριθμό πρέπει να αυξηθεί και να έχουμε παραγωγικέ και ανταγωνιστικέ επιχειρήσει. Ο πληθυσμό μα είναι κινητό και καλά ενημερωμένο, αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα να υπάρχουν και πολιτικέ που θα συνοδεύουν τα ωφέλη, όπω για παράδειγμα κατάρτιση έρευνα και ανάπτυξη. Τέλος, ευθύνη σημαίνει συνεργασία. Ε, κυρίως συνεργασία σε τελωνιακό επίπεδο, διότι οι πιο αποτελεσματικές διαδικασίες θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν να καταπολεμήσουμε την ε, παραποίηση και να διευκολύνουμε τις αλλαγές. Ολοκληρώνω, συνάδελφοι, ελπίζοντας ε, το έγγραφο αυτό να το εκφράζει τις απόψεις όλων στο μεγαλύτερο δυνατόν. Πριν ε, συντάξω την έκθεση, είχα κάνει ένα πρώτο γύρο διαβουλεύσεων σε διμερές επίπεδο και τώρα περιμένω και τη συνεισφορά σας εδώ στην Επιτροπή και μέσω τροπολογιών. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ την εισηγήτρια. Οι πολιτικές ομάδες τώρα. Θα ήθελα, επειδή το Μάιο θα έχουμε τη δυνατότητα να ξανασυζητήσουμε τις τροπολογίες, παρακαλώ τις πολιτικές ομάδες ε, να μιλήσουν, ε, αν το δέχονται, δύο λεπτά. Ο κύριος Κασπάρ για το ΕΛΚ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ πολύ την ε, συνάδελφο εισηγήτρια. Πολύ καλή και αντικειμενική σε μεγάλο βαθμό πιστεύω έκθεση. Ευχαριστώ πολύ γιατί ήδη στην έκθεση της ανέφερε σημεία τα οποία τα τελευταία χρόνια πάντα θεωρούσε σημαντικά το ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ επίσης για τις επικρίσεις ε, που εκφράζει έναντι της Κομισιόν με βάση αυτά τα οποία έχουμε ζητήσει και δεν έχει ακόμη ε, δεχθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προσβλέπω στην ε, καλή συνεργασία της επόμενης εβδομάδας όταν θα έχουμε και το κείμενο των τροπολογιών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. Σοσιαλιστές τώρα. Ο David Μάτσιν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τα 30 δευτερόλεπτα που με έδωσε ο συνάδελφος Κασπάρη. Θα είμαι συνοπτικός. Ευχαριστώ την κυρία Μπεγκίν για τη συνεργασία που είχαμε που ήταν θαυμάσια. Η έκθεσή της είναι μια πολύ καλή αφετηρία. Θέλω να τονίσουμε ότι η ομάδα μας εξακολουθεί να στηρίζει με κάθε αποφασιστικότητα το πολυμερές ε, εμπορικό σύστημα και στηρίζουμε τις διαπραγματεύσεις της ΝΤΟΑ Επίσης, θέλουμε να είναι εφαρμόσιμες ε, οι συμφωνίες από πλευράς συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών, περιβαλλοντικής βιωσιμότητας ε, και κοινωνικής υπευθυνότητα μπορούμε να ακολουθήσουμε τα παραδείγματα TTIP και TISA και σε άλλες ε, διαπραγματεύσεις για εμπορικές συμφωνίες. Θεωρούμε ότι η Επιτροπή πρέπει να κάνει περισσότερα για να παρακολουθεί την εφαρμογή και να εμπλέκει περισσότερο και το Κοινοβούλιο στην εφαρμογή των υπαρχουσών συμφωνιών ελευθερών Όσον αφορά τις ε, παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, είναι ουσιώδες στοιχεία λόγω της παγκοσμιοποίησης μας δίνουν τη δυνατότητα να υπάρξουν ε, θέσεις εργασίας ε, και καλές περιβαλλοντικές και κοινωνικές προδιαγραφές και βεβαίως και για τα ορυκτά από περιοχές συγκρούσεων πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι δεσμευτική η προσέγγιση τι δεν έχει καλύψει η ανακοίνωση της Επιτροπής. Για παράδειγμα δεν λέει τίποτα για την Κίνα και για το οικονομικό καθεστώς ε, αγοράς, το καθεστώς οικονομίας της αγοράς δηλαδή για την Κίνα. Πιστεύουμε ότι επίσης και οι εμπορικές ανταλλαγές πρέπει να επανεξεταστούν. Μας ε, απογοητεύει επίσης που δεν λέγεται τίποτα για το καθεστώς μετά ε, τη Συμφωνία Κοτονού. Πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό και δεν αντιμετωπίζει και μερικά από τα ευρύτερα θέματα που δεν είναι τόσο κεντρικά, αλλά που ίσως θα πρέπει να γίνουν κεντρικά, ιδιαίτερα ισότητα των φύλων μέσω της εμπορικής πολιτικής. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. ECR. Έμα Μακλάκη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι και εγώ όσο πιο σύντομη γίνεται. Να ευχαριστήσω και εγώ την εισηγήτρια που ήταν ανοιχτή και δεκτική για τροπολογίες, θα καταθέσουμε αρκετές. Εν γέννη θα πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο στις ευκαιρίες που προκύπτουν για πιο ανοιχτό εμπόριο. Τι μπορούμε να πετύχουμε μειώνοντας τους δασμούς, ε, καταργώντας τα μη δασμολογικά εμπόδια, βελτιώνοντας την κανονιστική συνεργασία κλπ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες και τις μικρές επιχειρήσεις που θέλουν να αυξήσουν τις εξαγωγές τους. Και όλα αυτά για να αυξήσουμε τις, ε, την απασχόληση και την ανάπτυξη. Πρέπει να δούμε ποιε είναι οι προτεραιότητές μα. και τι πρέπει να κάνει η Κομισιόν καλύτερα σε σχέση με το παρελθόν για να προχωρήσουμε σε διαπραγματεύσει που έχουν ξεκινήσει με την Ιαπωνία και τις ΗΠΑ για παράδειγμα. Πού θέλουμε να φτάσουμε και ελπίζουμε ότι θα ε, ξεκινήσουμε διαπραγματεύσει και με άλλε χώρε. τη Ασία. Επίσης θα πρέπει να εστιάσουμε στις ψηφιακέ υπηρεσίε, Σημαντικό κεφάλαιο για μας. Θα, κάνουμε, θα υποβάλουμε τροπολογίες και γι' αυτό. Ε, διαπραγματεύσεις που έχουν ολοκληρωθεί, επίσης θέλουμε να αναφερθούμε σε αυτές και στην εφαρμογή τους, ε, για παράδειγμα τη Σιγκαπούρη. Θα πρέπει εμείς να λάβουμε θέση, να τοποθετηθούμε ε, και αφού το συζητήσουμε για το παράνομο εμπόριο σε προϊόντα που έχουν σχέση με τη χλωρίδα και την, ε, με την πανίδα, άγρια πανίδα. Θέλουμε να υποβάλουμε και εκεί μια ε, τροπολογία. Γενικά θέλουμε να γίνει πιο φιλόδοξο, πιο θετικό το κείμενο ε, και να στηριχθεί από όλε ομάδε για να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα στην Κομισιόν. Ευχαριστώ. Για τους φιλελεύθερους ε, οι θετικές πτυχές είναι πολύ περισσότερες από τις αρνητικές ε, και αυτό θα πρέπει να είναι το βασικό μήνυμα της έκθεσής μας. Ε, καλωσορίζω το πρώτο κείμενο, το προσχέδιο και θα συνεργαστούμε για να έχει θετικό πρόσημο η τελική έκθεση. Η έκθεση αυτή είναι καινοτόμος, ε, βλέπει προς το μέλλον και αυτό θα πρέπει να είναι το τελικό αποτέλεσμα. Η προτεραιότητά μας είναι η ψηφιακή διάσταση του διεθνούς εμπορίου, η διευκόλυνση της ανταλλαγής ε, της, πρόοδου στον τομέα των υπηρεσιών και γενικότερα συμφωνίες 21ου αιώνα. Συνολικά μπορούμε να δουλέψουμε το προσχέδιο για να γίνει πιο ισορροπημένο Ε, πρέπει να στηρίξουμε και την επαναβιομηχάνηση της Ευρώπης αλλά και νέους τεχνολογικούς τομείς. Ε, προδιαγραφές, κανόνες είναι σημαντικοί αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα να δώσουμε βάρος και στους πολυμερείς κανόνες. Σε ό,τι αφορά το, στάτους, το καθεστώς αγορές για την Κίνα είναι σημαντικό να αναφερθεί αλλά γνωρίζουμε ότι υπάρχουν θέματα τα οποία θα πρέπει να λυθούν μέχρι το τέλο του χρόνου. Αυτό είναι ένα θέμα μάλλον που θα πρέπει να λυθεί μέχρι το τέλο του χρόνου, ενώ η στρατηγική αυτή είναι μακρόπνοη. Ξεπερνά την Κίνα. Επίση, θα πρέπει να πούμε περισσότερα για τι διαπραγματεύσει για την TTIP. Στο τελευταίο μα ε, ε, ψήφισμα ε, ζητήσαμε να ολοκληρωθούν επιτυχώ διαπραγματεύσει, ότι είναι σημαντικό πολιτικό σημείο αυτό. Επίση, χαίρομαι που δίδεται έμφαση στο ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, επιχειρήσεων στο διεθνέ εμπόριο και θα υποβάλουμε και κάποιε τροπολογίε. Ευχαριστώ. Helmut Scholz. Α, όχι. Ποιο. Α, ο κύριο Σόλτ. Να ευχαριστήσω και εγώ την εισηγήτρια. Νομίζω ότι αναφέρθηκε πολύ αναλυτικά στις διάφορες πλευρές του θέματος. Ε, θέλουμε δίκαιο εμπόριο. Αυτό είναι καινοτομία στην ε, εμπορική στρατηγική της Κομισιόν. Πρέπει να το τονίσουμε περισσότερο. Ούτω ώστε να υποχρεωθεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λαμβάνει υπόψη αυτό το θέμα στις εμπορικές και οικονομικές διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για το πόσο συγκεκριμένη είναι και πόσο συγκεκριμένα παραδείγματα θέτει για τις διάφορες προκλήσεις. Οπωσδήποτε θα υποβάλουμε τροπολογίες όπου θα επιχειρήσουμε είτε να εμβαθύνουμε ή να σταθμίσουμε διαφορετικά διάφορα θέματα. Και στο τμήμα όπου λέμε ότι πρέπει να καθορίσουμε την εμπορική μας στρατηγική σε σχέση με τις πολυμερείς διαπραγματεύσεις ε, που διεξάγει η Ένωση. Θέλουμε εκεί να ληφθεί υπόψη η δημογραφική εξέλιξη. Το 2050 η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει το πολύ 480 εκατομμύρια, ενώ η Αφρική θα έχει 2,3 έως 2,4 δις η Ασία, η Λατινική Αμερική, πολύ κόσμο. Άρα θα έχουμε άλλες εμπορικές ε, ροές από αυτές ε, που έχουμε τώρα. Πρέπει λοιπόν να τις λάβουμε υπόψη τώρα που σχεδιάζουμε την ε, μελλοντική μας εμπορική στρατηγική και για την Κίνα. Βεβαίως πρέπει να πούμε πράγματα πιο συγκεκριμένα. Αλλά το καθεστώς οικονομίας της αγοράς είναι ένα πολύ μικρό τμήμα του διακυβεύματος. Πρόκειται για τεράστια αγορά πώς θα χειριστούμε μια τέτοια τεράστια αγορά από πλευράς ε, συνεργασίας για το εμπόριο και την οικονομία. Και κάτι άλλο. Συζητήσαμε μόλις προηγουμένως τον προϋπολογισμό. Να σκεφτούμε, πιστεύω, σε βάθος, να ξανασκεφτούμε σε βάθος τον προϋπολογισμό μας σε σχέση ακριβώς με την εμπορική πολιτική της Ένωσης. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ, Χέλμουτ. Λοιπόν, έχουμε υπερβεί το χρόνο, παίζουμε ήδη τις καθυστερήσεις. Να δώσω το λόγο στη ΣΚΑ. Ευχαριστώ. Αντικαθιστώ τον συνάδελφο που δυστυχώς δεν μπορεί να είναι εδώ. Δεν μπορώ βέβαια να τη συνοψίσω τις σημειώσεις του τόσο γρήγορα. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, αυτό είναι βέβαιο, και σίγουρα θα υποβάλουμε και τροπολογίε ως προς την ανάγκη να αλλάξει λίγο η νοοτροπία, γιατί δεν θεωρούμε ότι θα λύσει τα εσωτερικά μας προβλήματα η εμπορική πολιτική. Μπορούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα σε θέματα διαφάνειας και δημοκρατίας, ε, βιώσιμες παγκόσμιες αλυσίδες αξιών. Εδώ μπορούμε να έχουμε αποτελεσματικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι αλυσίδες αξιών θα ε, είναι κάτι που θα διαχειριζόμαστε υπεύθυνα. Και επίσης ένα πολύ σημαντικό είναι ε, η πολυμορφία. Δεν θα πρέπει να αποφύγουμε αυτή την πολυμορφία. Θα πρέπει ο ΠΟΕ να βρίσκεται στο επίκεντρο των στρατηγικής μας. Αυτά λοιπόν ήταν ε, η, η πολύ σύντομη περίληψη προς την κατεύθυνση των τροπολογιών μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ένα μέλος έχει ζητήσει τον άδελφο, ο συνάδελφος Μορέλ, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται πράγματι για μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση, η οποία θα πρέπει να αποτελέσει κίνητρο για μα ε, μέλη τη Επιτροπής Εμπορίου να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει μια διανοητική επανάσταση σε θέματα ε, Ευρωπα... εμπορίου. Θα μπορούσαμε να πούμε, είπε πολύ συχνά και η συγκήτρια, ότι τα συνήθεια, αλλά πολύ σωστά είπε η συγκήτρια πρέπει να συμμετέχουν και οι πολίτε με πλήρη διαφάνεια για τι εμπορικέ συμφωνίε και αυτό το μήνυμα πρέπει να περάσει. Η κυρία Μάλστρομ από αυτή την άποψη έκανε κάποια πρόοδο σχέση με τον προκάτοχό τη, αλλά έχουμε πολύ δρόμο ακόμα προκειμένου να περάσουμε από τα λόγια στι πράξει και να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτό το οποίο αποκαλούμε εμεί τι δίκαιε ανταλλαγέ, δηλαδή όχι τη θρησκεία των ελεύθερων ανταλλαγών, αλλά κατάλληλου κανόνε. Θα ήθελα να σταθώ σε τρία σημεία στις προτάσεις της Επιτρόπου πολύ συχνά ξεχνάμε κάποια πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Γεωργία και βιομηχανία. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Στην TTIP, στη ΣΕΤΑ, στο Μερκοσούρ, στην Αυστραλία, στη Νέα Ζηλανδία. Θα πρέπει να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιδείξει σοφροσύνη, διότι διαχειρίζεται ευαίσθητα γεωργικά προϊόντα. Παραδείγματο χάρη, βόηο κρέα, ε, χείριο κρέα. Θα πρέπει ε, επίση να ξαναδούμε το θέμα του ε, καθεστώτο οικονομία τη αγορά τη Κίνα πιέζει ο χρόνος και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να λάβει σαφή θέση. Δεν πρέπει να υπάρχουν άλλε αμφισημίε, έχουμε αρκετέ. Και ένα τρίτο, αυτό δεν δεσμεύει την ομάδα μου, για το θέμα της πρόσβασης στι ε, δημόσιε αγορέ. Αυτό θα γίνει όλο ένα και πιο σημαντικό και κάποια στιγμή, εάν οι εταίροι μας δεν συμφωνούν να ανοίξουν τις δημόσιες αγορές τους, εμείς ως Ευρωπαίοι θα πρέπει να επιδείξουμε την ευφυΐα να σκεφτούμε κι εμείς ε, μιας, ε, ε, την ιδέα μιας ευρωπαϊκής πράξης. Νομίζω ότι επί τη ευκαιρία αυτής της έκθεσης θα μπορέσουμε να εμβαθύνουμε στις συζητήσεις που ενδιαφέρουν το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφε και τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τη Γενική Διεύθυνση Trade ο Ιαν Φόλμπραχτ, ε, έχετε το λόγο, ε, πρέπει να είστε σύντομοι. Αναφερόμαστε επανάσταση μένα, αλλά σύντομα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, εξότιμα μέλη. Ευχαριστώ. Αν μου επιτρέψετε, σε 1,5 λεπτό δεν μπορώ να ανατρέψω τα πάντα, αλλά θα κάνω ό,τι μπορώ. Ευχαριστώ την κυρία Μπέγκιν και τους συναδέλφους της. Είχα την ευκαιρία να τη γνωρίσω να ασχοληθώ με ορισμένα μόνο, δεν μπορώ να καλάψω τα πάντα για τη διαφάνεια. Έχουμε κάνει ουσιώδεις προσπάθειες τα τελευταία χρόνια και ήταν ε, βασική εστίαση της στρατηγικής μας για το εμπόριο. Σχετίζεται και με κάτι που είπε ο κύριος Μάρτιν. Δημοσιεύουμε τις διαπραγματικές εντολές, τις προτάσεις ε, για διαπραγματεύσεις, ε, διάλογος με την κοινωνία των πολιτών. Αν τα δείτε αυτά σε σχέση με πώ ήταν τα πράγματα πριν από 10-15 χρόνια όταν είχαμε τι διαπραγματεύσει στο Κανκούν και στο Χονγκ Κονγκ ε, ήταν πολύ διαφορετική κατάσταση. Έχει υπάρξει μεγάλη πρόοδο, πιστεύω. Και αυτό έγινε και επειδή ακούσαμε αυτά που λένε οι συνάδελφοι εδώ για την ισότητα των φίλων. απαντώντα τον κύριο Μάρτιν, βεβαίω το λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη, για την ΤΙΣΑ θα μεταφέρω στον συνάδελφο που ασχολείται για τα θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς σημειώνουμε και, και καλωσορίζουμε την έμφαση του Κοινοβουλίου γι' αυτό, αν μπορούμε να επιτύχουμε αποτελέσματα για όλα, είναι συζητήσιμο, αλλά χαιρόμαστε για αυτή τη νέα έμφαση. Για τον κύριο Κασπάρη θα περιμένουμε τις τροπολογίες του. Τον ευχαριστούμε για, τις, ε, για τα θετικά σχόλια, για τα σχόλια του κύριου Μάρτιν, για το πολυμερές σύστημα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε είναι αλήθεια, σχετίζεται και με κάτι που είπε η κυρία Κέλλερ αυτό, για τον τρόπο εφαρμογής και την αξιολόγηση της εφαρμογής βεβαίως είναι βασικό. Ίσως μας χρειάζεται λίγος χρόνος και εντός της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου για να σημειώσουμε πρόοδο, αλλά προσπαθούμε. Για το καθεστώς ε, της Κίνας συζητείται σε τόσο πολιτικό επίπεδο, σε τόσο υψηλά πολιτικό επίπεδο, που ε, καλύτερα να μας τα πει η κυρία Μάλστρομ. Αλλά βεβαίως εμείς σε επίπεδο υπηρεσιών το γνωρίζουμε. Η κυρία Μακλάρκιν ε, αναφέρθηκε στις ψηφιακές υπηρεσίες στη Γενέβη. Αυτή τη στιγμή στα πλαίσια της κατάστασης μετά από τον Αϊρόμπι βεβαίως και μας απασχολεί. έθιγε επίσης ε, το θέμα ότι τα θετικά είναι περισσότερα από τα αρνητικά και ελπίζω αυτή η προσέγγιση να γίνει ακόμη πιο θετική στην έκθεση μέσω τροπολογιών. Δεν υποτιμούμε τη σημασία των αρνητικών επιπτώσεων όπου προκύπτουν, αλλά νομίζω ότι πολλά μέλη της Επιτροπής θα θεωρούσαν, όπως λέει και η Επιτροπή, ότι ο λόγος για τον οποίο θέλουμε να έχουμε ευρείες και συνολικές συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου είναι ότι, ότι με αυτόν τον τρόπο έχουμε περισσότερα θετικά από ότι τα αρνητικά. Ελπίζω να μας στηρίξετε σε αυτό. Σημείωσα τα σχόλια του κυρίου Σόλτς για τις δημογραφικές εξελίξεις. Εντάξει, νομίζω ότι δεν ε, ανέτρεψα τα πάντα και ευχαριστώ για την υπομονή σας. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Η συγκήτρια έχει σχόλια, αν χρειάζονται, σύντομα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε επειδή δεν έχουμε και χρόνο, να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους ε, για τη συνεισφορά τους και ε, για την ευελιξία που επέδειξαν. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε μια βαθύτερη συνεργασία στις επόμενες συναντήσεις και ελπίζω στην επόμενη συζήτηση που θα γίνει εδώ στην Επιτροπή μας θα έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο ίσως για αυτή τη συζήτηση, η οποία σίγουρα απαιτεί ε, ένα πιο ευέλικτο ε, πρόγραμμα. Ευχαριστώ πολύ. Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών 25 Απριλίου, 12 το μεσημέρι. Πέρα τη συνεδρίαση, να σας πω ότι στις 3 το απόγευμα θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας και θα είναι εδώ η Υπουργό ε, Διεθνούς Εμπορίου του Καναδά, η Κρίστια Φρίλαντ. Ε, ευχαριστώ. Και ο Πρόεδρος ευχαριστεί και τους διερμηνείς.